του Κοινοβουλίου, οι δε τίτλοι αυτών των ε, πράξεων πρόκειται να μνημονηθούν ή στα πρακτικά. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ελάβαμε έναν κατάλογο με κάποιε προτάσει για ορισμό κάποιων μελών για αντιπροσωπείε, αλλά και ε, επιτροπέ και αντιπροσωπείε. Όλα αυτά δημιουργούν στα ε, ε, πρακτικά εφόσον ε, δεν υπάρχει απιένσεις θα εγκριθούν οι τοποθετήσει αυτών των συναδέλφων. Προχωρούμε τώρα. Σύμφωνα με την